Ladies and gentlemen, we have to get... Καλημέρα σας. Πρέπει να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Είναι 10 και 10. Σας παρακαλώ πολύ όλους να καθίσετε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε μια μικρή καθυστήρηση. Πολλά μας έχουν μείνει. Στις 11 και 4 θα αφήσω την Προεδρία γιατί πρέπει να πάω στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκεί να πω δύο λόγια. Θα δούμε όμως ποιο ε, ποιος θα βρεθεί στην Προεδρία. Ε, τρεις διαφορετικοί πρόεδροι, ποιος τη χάρη σας. Να περάσουμε λοιπόν στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης, να προτείνω να την εγκρίνουμε. Ωραία. Δύο. Πρακτικά. Σας έχουν μοιραστεί. Εάν υπάρχουν σχόλια, παρακαλώ πολύ μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να μας το πείτε. Διαφορετικά θα θεωρούνται εγκεκριμένα. Ανακοινώσεις του Προέδρου. 21 Νοεμβρίου μας έστειλε τη θέση μας για τον προτινόμενο κανονισμό για την, ε, τα περιπτώμενα αλλιεύματα και το μήνυμα ε, μαζί τη μια συζήτηση. Εμείς στις 16 Απριλίου στην Ολομέλεια εγκρίναμε το ψηφίσμα για να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και τότε είπα ε, διαπραγματευτική εντολή η οποία στη συνεδρία αυτή θα πρέπει να εγκριθεί. Να σας πω πως η νέα συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικής ε, τεχνολογίας έχει ξεκινήσει. Αυτά τα e-meeting λοιπόν θα γίνονται, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα tablet και, για, και τα τηλέφωνά μας και θα έχετε και πια με αυτόν τον τρόπο όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για τη δουλειά μας. Όπως επίσης και παρουσιάσεις που ε, θα βλέπουμε εμείς εδώ live. Μπορείτε λοιπόν να είσαστε σε άμεση επαφή μαζί μας και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε και για επικοινωνία με το προσωπικό σας. Έτσι λοιπόν δεν θα εκτυπώνουμε και τα έγγραφα των ε, συνεδριάσεων και πολλές επιτροπές έχουν περικόψει κατά 40% το χαρτί που καταναλώνουν. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, το e-meeting, και να βελτιστοποιήσετε την, τον αντίκτυπο που θα έχει στην εξοικονόμηση ε, πόρων. Τώρα, για την ακρόαση που θα γίνει 16 Δεκεμβρίου για την Μεσόγειο, όλα τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα αρκετές μέρες πριν την ε, ακρόαση αυτή. Χαιρετίζω λοιπόν το ότι θα γίνονται αυτές οι συνεδριάσεις ηλεκτρονικά. Πάντως η αλήθεια είναι πως κάποιος έκανε hacking στο, στην υπηρεσία Wi-Fi του Κοινοβουλίου και όπως θα καταλάβατε δεν έχουμε πλέον δίκτυο. Οπότε στο Info Center όπου χρειάζεται κανείς το ε, πιστοποιητικό που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στο Wi-Fi, οι ουρές είναι τεράστιες Άρα λοιπόν η πραγματικότητα αυτής της ηλεκτρονικής συνεδρίασης και η πόθη μας δεν συμπίπτουν απόλυτα. Ελπίζω πάντως πως Wi-Fi θα έχουμε σύντομα. Τώρα για τις ανακοινώσεις του Προέδρου υπάρχουν σχόλια, αν όχι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το 3. Για το ρόλο των γυναικών λοιπόν στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Η Ντολόρης Γκαρσία Γκέρο είναι η συγγήτρια. σοσιαλιστές 23 Απριλίου έλαβαν αυτή την γνωμοδότηση πρωτοβουλίας και έχουμε εδώ την συνάδελφο, την κυρία Γκαρσία Ιέρο, διορθώνω, η οποία είναι η η συγγήτρια. Έχουμε την Επιτροπή ΦΑΜ, η οποία ζήτησε να ισχύσει το άρθρο 51 του κανονισμού, να κάνουμε μια κοινή συνάντηση των δύο επιτροπών μας. Θα εφαρμοστεί λοιπόν, άρα Σήμερα μπορούμε να καλωσορίσουμε τα μέλη της Επιτροπής για την Ισότητα, για τις γυναίκες, συν εισηγητής είναι ο κύριος Ρωμέβα των Πρασίνων από τη δική τους επιτροπή που είναι και, δικός μας, ε, και δικό μας μέλος ο οποίος είναι καθοδόν. Φαντάζομαι πως σύντομα θα φτάσει. Στις 17 Ιουνίου κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και στις 14 Οκτωβρίου κάναμε και μια δημόσια ακρόαση με μεγάλο ακροατήριο. Οι ομιλητές σήμερα θα παρουσιάσουν το σχέδιο έκθεσης, θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και η ιδιομορφία της χρήσης του άρθρου 51 μας αναγκάζουν το να κάνουμε ένα μικρό αριθμό κοινών συνεδριάσεων. Σίγουρα θα εργαστούμε αποτελεσματικά και θα ξεπεράσουμε οποιασδήποτε διοικητικές δυσκολίες αντιμετωπίσουμε. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, να σας πω πως η καταληκτική ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες είναι 4 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Η κυρία Γκαρσία Ιέρο λοιπόν ως εισηγήτρια από την Επιτροπή μας έχει το λόγο. Ντολόρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με κάθε ηλεκτρίνεια γιατί εάν εσείς δεν είχατε δείξει αυτό το ανεξάντλητο πάθος για να συζητήσουμε και να καταθέσουμε την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Αλίας, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Ευχαριστώ λοιπόν τους υπαλλήλους μας που με τόσο ενδιαφέρον μου είπαν πως χρειάζεται ενημέρωση η πρόταση που χρονολογείται από το 2005 και η οποία αναγνωρίζει ποια είναι η έλλειψη ισότητας ή οι μειωμένες ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες που δουλεύουν στο χώρο της αλληλείας. Όχι μόνο στην αλληλεία, αλλά και στην εμπορία και στην μεταποίηση. Παρόλο που οι δύο αυτοί χώροι ρυθμίζονται από άλλες συλλογικέ συμβάσεις στα κράτη-μέλη με αποτέλεσμα εκεί τα προβλήματα να είναι μικρότητα εκεί τουλάχιστον εξασφαλίζονται κάποια ίσα δικαιώματα, αν όχι ίση μισθή. Όχι όμως στις γυναίκες που δουλεύουν πάνω στα σκάφη. Θέλω να ευχαριστήσω και τη βοηθό μου γιατί καταλαβαίνετε πως πριν μία έκθεση που αντικατοπτρίζει μία πραγματικότητα χρειάστηκε να γυρίσει όλα τα γραφεία του Κοινοβουλίου και να ψάξει πληροφορίες που θα επιτρέψει να καταθέσουμε αυτό το σύντομο σχέδιο. Γιατί δυστυχώς δεν είχαμε ούτε εκθέσεις, ούτε στατιστικά στοιχεία τα οποία από το 2005 και τα λοιπά να είχαν ε, συλλεχθεί. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους ε, συναδέλφους που τόσο με βοήθησαν. Το να λείπουν τα στατιστικά στοιχεία είναι ένα πρόβλημα που επιμένει και το οποίο δυσκολεύει ιδιαίτερα την κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης. Όταν θέλει κανείς δηλαδή να ποσοτικοποιήσει ε, την έλλειψη ισότητας, τις ανισότητες τις, ε, που προέρχονται από το φύλλο, ε, τις μισθολογικές ανισότητες, νομίζω πως Το βασικό ήταν η δέσμευση που αναλάβαμε και την οποία, στην οποία ανταποκριθήκαμε με την έκθεση αυτή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με τον κύριο Ρωμέβα. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και για το περιεχόμενο και σε προσωπικό επίπεδο και προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε όσο μπορούμε ε, όλους γύρω μας. Το λέω γιατί η πρωτοβουλία αυτή σε αυτό το χρόνο και κάτι που κοιτάμε τους διάφορους κανονισμούς, τους βασικούς κανονισμούς και άλλες προτάσεις, μας υπέδειξαν πως θα πρέπει να φανούν περισσότερο οι γυναίκες σε αυτό τον επαγγελματικό κλάδο και η συμβολή τους, γιατί σε κάποιες περιοχές και περιφέρειες της Ευρώπης δεν είναι μόνο μια παράδοση η συμμετοχή τους, δεν είναι μόνο πιο βιώσιμη η αλληλεία λόγω της συμμετοχής τους, αλλά είναι και το βασικό εισόδημα για τις ίδιες και για τις οικογένειές τους. Έτσι λοιπόν και στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς φαίνεται το θέμα της συμμετοχής γυναικών και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να προκρίνουν τη συμμετοχή τους στις ενώσεις παραγωγών, στις ενώσεις, α, των, ενώσεις στις συντεχνίες και να παρουσιάσουν μέτρα τα οποία κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον όσα έχουμε εδώ στο έγγραφο είναι μέτρα και τροπολογίες πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέροντα που επιτρέπουν και τη δημιουργία ενώσεις γυναικών έτσι ώστε να οργανωθούν καλύτερα όπως γίνεται από τότε που δημιουργήθηκε το δίκτυο γυναικών, η επαγγελματική κατάρτιση και κυρίως για τις νέες γυναίκες που εάν θέλουν ε, θα μπουν στον κλάδο με συνθήκες ισότητας. Και αυτό να γίνει με πληροφορίες στατιστικές που θα έχουμε, που θα μας επιτρέψει να κάνουμε μια κατανομή ανά τόπο, ανά ηλικία, ανά ποιος εργάζεται στον κλάδο, με τι μισθό και ποια είναι η επαγγελματική του κατάσταση. Στην έκθεση αυτή ζητήσαμε να αναγνωριστεί πως αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα που είναι μια οικονομική δραστηριότητα συγκεχημένη ενδεχομένως καμιά φορά ή μη αναγνωρισμένη, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και θα πρέπει να προστατεύεται και θα πρέπει να έχει κοινωνική κάλυψη, υγειονομική κάλυψη, σταξιοδοτική κάλυψη, παράλληλη με αυτή με αυτή που έχουν οι γυναίκες στην γεωργία. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιους διακρίσεις σε ένα χώρο στην Ευρώπη τον οποίο εμείς εκπροσωπούμε. Η οδηγία του 2010 για τους ελεύθερους επαγγελματία 2010 κάθετο 41 μας φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα γιατί θα επιτρέψει μέσα σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία που ζητήσαμε και τα οποία ζητήσαμε ανά περιφέρεια γιατί ενδιαφερθήκαμε κυρίως για τις γυναίκες που έχουν αναλάβει αυτό το έργο γιατί ξέρετε τι συμβαίνει σε συνθήκες κρίσης. Είναι κυρίως οι νέες γυναίκες οι οποίες χάνουν τη δουλειά τους. Δουλειές τις οποίες ασκούν κατά παράδοση και πολλές φορές έχει χρειαστεί να στραφούν σε νέες ε, ε, δραστηριότητες και ξέρετε πως αυτές τις στιγμές ασχολούνται και με την παράκτια αλληλεία αλλά πολλές φορές ασχολούνται και με την εκτροφή, με την υδατοκαλλιέργεια, μαζεύουν ε, μύδια, όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο ορατές, θα πρέπει η συμβολή τους στις ε, περιφέρειες που εργάζονται, στις ζώνες που εργάζονται, να αναγράφεται στα στατιστικά δεδομένα που συλλέγουμε. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάτι που ακούστηκε στην ακρόαση. Υπάρχουν και συγκεκριμένες ασθένειες ε, που πλήττουν αυτό το επάγγελμα. Και αυτό είναι μια παλιά διεκδίκηση της ε, συναδέλφου εδώ στην Επιτροπή και θεωρούμε πως θα ήταν δίκαιο αυτές οι ασθένειες που αποτελούν συνέπεια συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας να εμφανίζονται και να θεραπεύονται από τα συστήματα υγείας και περίθαλψης κάθε κράτους μέλους. Έχουμε μια σειρά μέτρα σημαντικά που έχουν να κάνουν με την ε, συμμόρφωση με το σχέδιο για τις ίσες ευκαιρίες που εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο και όπου θα πρέπει να συμφιλιώνεται αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα με την οικογενειακή και την ιδιωτική, την προσωπική ζωή. Στην ε, έκθεση του 2005 μιλούσαμε για γυναίκα και οικογενειακό εισόδημα, κάτι το οποίο πια δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Γιατί αν το δούμε έτσι δεν ζούμε σε συνθήκες ισότητας. Γιατί αν οι γυναίκες δεν αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στην οικονομία είτε την επίσημη είτε τη μαύρη, ε, το κατά πόσο το εισόδημα το οποίο κερδίζουμε είναι για την οικογένειά μας ή για εμάς δεν θα έπρεπε να έχει σημασία. Και αυτό εμφανίζεται και στην έκθεση τη σημερινή. Θα πρέπει δηλαδή πια στον 21ο αιώνα να γνωρίζουμε πως κάποιες γυναίκες ασκούν αυτή τη δραστηριότητα που θα πρέπει να αναγνωρίζεται και που να έχει ε, δικαιώματα να την ασκούν για τους δικούς τους λόγους για να επιβιώσουν οι ίδιες. 100.000 γυναίκες εμπλέκονται σε όλη την Ευρώπη στο θέμα αυτό περίπου γιατί όπως είπα τα στατιστικά στοιχεία εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να τα επικυρώσουν και θα πρέπει να επαγρυπνούν έτσι ώστε να συμμορφωθούν με την οδηγία στην οποία αναφέρθηκα. Στο διάστημα αυτό λοιπόν που συζητάμε τους κανονισμούς φαίνεται πως οι γυναίκες μέσω των ε, ευρωβουλευτών αισθάνθηκαν πως ε, αυτά τα οποία είχαμε εδώ ή τα όσα είχαμε στην έκθεση Φερέιρα, οι διάφορες τροπολογίες, δεν διατηρήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι καλό που η έκθεση αυτή έτσι εμφανίζεται τώρα εκ των υστέρων έτσι ώστε και η Επιτροπή και το Συμβούλιο να ευαισθητοποιηθούν και να εντάξουν αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω δεν, εντάχθηκαν, δεν, έγιναν, δεν εγκρίθηκαν στις τροπολογίες μέσω της δικής μας έκθεσης και να αναγνωρίσουν αυτή την πραγματικότητα, να πούνε πως η ισότητα στις ευκαιρίες και η αναγνώριση είναι πλεονέκτημα και για τις ίδιες τις κοινότητες τις οποίες διαβιώνουν οι γυναίκες αυτές. Γιατί έτσι και εμείς αισθανόμαστε πως αποτελούμε τμήμα της ευημερία και της οικονομικής και της ε, πολιτιστικής και της ε, περιβαντολογικής βιωσιμότητας της ε, κοινωνίας μας. Και βεβαίως έχουμε πολλές εμπειρίες να μεταδώσουμε σε παιδιά, σε συντρόφους και μπορεί να αποτελέσουν και νέες πηγές Σε κάποιες περιφέρειες δε, και το γνωρίζω αυτό, έχουν ως σκοπό να συνδυάσουν την αλληλεία με ε, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό έτσι ώστε να αναζωπυρώσουν τις περιοχές αυτές οι οποίες πραγματικά βρίσκονται σε παρακμή. Θα πρέπει λοιπόν να εντάξουμε ε, αυτά τα οποία άπτονται της επαγγελματικής ζωής των γυναικών σε αυτόν τον κλάδο και να αναγνωρίζεται μια και καλή ο ρόλος τους, να είναι πια ορατές. Έκανα προσπάθεια, όπως έκαναν και οι υπηρεσίες της Επιτροπής και ο συνάδελφος, να εντάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία διάφοροι συνάδελφοι μας ζήτησαν. Είναι θετικά για να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά είμαι ανοιχτή το είπα την πρώτη φορά που πήρα το λόγο σε οποιαδήποτε πρόταση την οποία εσείς θα καταθέσετε και που θα βελτιώσει την έκθεσή μας. Και θα τη συμπληρώσει. Γιατί σίγουρα κάτι μας ξέφυγε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much indeed, uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρστία Ιερό, για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει στην έκθεση. Το εκτιμούμε πολύ αυτό. Επίσης να πω ότι σήμερα έχουμε την ε, τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Γιαρόκα και τον κύριο Ρωμεύα, ο οποίος μόλις έφτασε. Κυρία Γιαρόκα, θα θέλατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Για εμάς, αυτός ο τομέας ήταν πάρα πολύ σημαντικός για εμάς, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε, που εξηγούν γιατί πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το ζήτημα. Ένας από τους λόγους είναι η διαχείριση της ε, κρίσης και το πώς συνδέεται η φτώχεια με τις ε, συνθήκες διαβίωσης αυτών των γυναικών. Και είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το πώς αυτό συνδέεται με τον ε, αλλιευτικό τομέα και το μέλλον αυτού, το πώς η φτώχεια μπορεί να καταπολεμηθεί μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικά και οικονομικά, με δημιουργία καλύτερων θέσεων απασχόλησης όταν ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό μάλλον να υπάρξει βελτίωση, γι' αυτό και εμείς στηρίζουμε ευθύ εξ αρχής αυτήν την ε, έκθεση. Επιπλέον, οι δυνατότητες που ε, έχουν γυναίκες για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά πρέπει να αυξηθούν όχι μόνο ε, σε, στα κέντρα αλλά και στις ε, ακτές και στις παράκτιες περιοχές όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για θέσεις εργασίας. Ξέρω πως ε, έχετε περιορισμένο χώρο στην εκθεσή σας, περιορισμένο αριθμό λέξεων, αλλά ε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε και το ρόλο των γυναικών αυτών ε, ως ε, μέλη οικογένειας. Εμείς ε, λοιπόν θα ενισχύσουμε τις προτάσεις σας για δημιουργία περισσότερων επενδύσεων έτσι ώστε οι γυναίκες να βελτιώσουν τις ε, συνθήκες διαβίωσής τους και ε, τις συνθήκες απασχόλησής τους στον τομέα της αλληλείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γιαρόκα. Ο κύριος ε, Ρωμέβα τώρα πρόλαβε να έρθει. Είναι ο συνεισηγητής της δική μας επιτροπής και του δίνω μέσω στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την αργοπορία μου. Μόλις έφτασα από την Νότια Αφρική, ε, ήμουν στη συνεδρίαση ΆΕΚΑΤ και τελείωσε προχθές, όμως το αεροπλάνο μου πέταξε χθε, γι' αυτό και άργησα. Είχα μια μικρή καθυστέρηση. Γνωρίζω ότι η κυρία Γκαρσία ήδη σα έχει ενημερώσει για το περιεχόμενο της έκθεσης. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τονίσω δύο-τρει επιτυχίες που θεωρώ πολύ σημαντικές. Γιατί η έκθεση αυτή είναι σημαντική και γιατί εγώ ήθελα προσωπικά να συμμετέχω σε αυτή την έκθεση. Παρακολούθησα πολλές περιπτώσει, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και στη χώρα των Βάσκων και σε άλλες περιοχέ όπου παρατηρήθηκαν ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες, στι οποίε στις οποίες εργάζονταν οι γυναίκες στον χώρο της Αλία. Οι γυναίκες αυτές δεν φαίνονται καθόλου, να πω. Και πρέπει να φέρουμε στο φως και να τονίσουμε τον ρόλο των γυναικών στον αλλιευτικό τομέα. Γνωρίζουμε ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα μια τέτοια έκθεση, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να ε, αναγνωρίζουμε το ρόλο μας ως θεσμικό όργανο στην προσπάθεια αναγνώρισης του ρόλου των ε, γυναικών στον αλλιευτικό τομέα. Και όχι μόνο ότι το ρόλο τους αλλά και τις συνέπειες που έχει αυτό, νομικές, ε, συνέπειες ασφάλισης. Έπειτα, θεωρώ επίσης σημαντικό ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το ρόλο των γυναικών στην Αλία. Για πάρα πολύ καιρό οι γυναίκες και ο ρόλος τους στην Αλία ήταν άμεσα συνδεδεμένος με, τον, ε, ε, το επάγγελμα των συζύγων τους ή των γονιών τους, των ανδρών. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε τις ε, γυναίκες από τους άνδρες στην Αλία, να τις δούμε ως ε, μεμονωμένες ε, προσωπικότητες και με αυτόν τον τρόπο να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα του παρελθόντος. Μία ευκαιρία να το κάνουμε αυτό είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένας άλλος τρόπος είναι η εφαρμογή της νέας ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής και πιστεύω πως αυτό, αυτή η πολιτική είναι κάτι που μπορεί να επιδεχτεί πολλές βελτιώσεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Γκαρσία Ιέρο για την δουλειά που έκανε. Εκτιμώ όχι μόνο την ε, πολλή δουλειά που εκείνη και η ομάδα της έκανε, αλλά και το ότι δεν ήταν, δεν ήταν και εύκολο το έργο. Ωστόσο, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της και ήταν πολύ εύκολο να οδηγηθούμε σε συνένεση. Και πραγματικά είναι ένας ε, τομέας τον οποίο πρέπει να ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και ξανά ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε εσεί για την έκθεση αυτή και ξέρω ότι και εσεί και η κυρία Φράγα μόλι ήρθατε από την Νότια Αφρική. Ελπίζω να μην είστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Έχω τώρα ένα κατάλογο μιλητών, καταρχήν η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Δολόρης Γκαρσία και τον κύριο Ρωμέβα για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Και όπως ε, παρουσιάστηκαν ε, κάποιες ε, τροπολογίες σε άλλες περιπτώσεις για την μεταρρύθμιση τη συνεθνική πολιτική. Εγώ αισθάνομαι σήμερα ότι αποτείω από το φόρο τιμή σε πολλέ γυναίκε, όπω στη γιαγιάδε μου και στη μητέρα μου, που συνέβαλαν στο να μπορούν να φύγουν τα σκάφη, να ετοιμάζουν το φαγητό, να είναι τα δίχτυα έτοιμα οποιαδήποτε στιγμή. Όλες αυτές είναι αόρατες ιστορίες. Γι' αυτό το πρώτο που θέλω να τονίσω στην έκθεση αυτή είναι ότι αποτελεί ένα βήμα για να καταστήσει ορατό το ρόλο των γυναικών και περισσότερο για το μέλλον θα έλεγα Ορισμένοι από εμά ε, θυμούνται συναισθηματικά και το παρελθόν και θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ε, για τους ανθρώπους της θάλασσας. Επίσης, αξιολογώ θετικά την αναγκαιότητα να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις ε, της δουλειάς των γυναικών στη θάλασσα, να, κάνουμε, λοιπόν, να χαράξουμε κάποιες στατιστικές και να δούμε ποιες διάφορες καταστάσεις υπάρχουν σε κάθε μία περιφέρεια και σε κάθε μία χώρα για το θέμα αυτό. Εμείς ε, αναφερθήκαμε στην αναγκαιότητα αναγνώρισης των νόσων, των επαγγελματικών νόσων. Δυστυχώς δεν υπάρχει ενερμόνιση στην νομοθεσία των κρατών μελών. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό θέμα της κατάρτιση των γυναικών που τώρα ασχολούνται με την αλία και επίσης είναι σημαντική και η κατάρτιση των γυναικών οι οποίες στις ζώνες όπου θα υπάρχει σοβαρή αναδιάρθρωση θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα, θα πρέπει να βρουν νέες θέσεις εργασία και νέου τρόπου εργασία που μπορεί να συνδέονται με τη θάλασσα έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα της κατάρτισης, της επαγγελματική ε, διαφοροποίησης και τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε και τους πιο νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το ρόλο των γυναικών, όπως είδαμε και στην ακρόαση εδώ στο Κοινοβούλιο. Και έχουμε δύο προκλήσεις ενώπιον της αποτυχίας και της προσπάθειας που κάναμε με διάφορες τροπολογίες για να δώσουμε και μία προοπτική φύλου στην ε, αλληλευτική πολιτική, όπως κάναμε με το πρόγραμμα Ορίζοντας. Στην περίπτωση αυτή αποτύχαμε γιατί δεν κατορθώσαμε να συμπεριληφθεί αυτή η προοπτική του φύλου. Επομένως, η πρόκληση που έχουμε στην έκθεση αυτή είναι να κάνουμε μια σωστή διάκριση σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ποιες είναι οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμών και ποιες οι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και σαφήνεια για να μην δημιουργήσουμε σύγχυση στον κλάδο και στις γυναίκες που αυτή τη στιγμή δίνουν πολύ μεγάλη προσοχή και στη δουλειά που κάνουμε εμείς στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, από κοινού πρέπει να κάνουμε αυτή την πορεία, αλλά διαβάζοντα και την έκθεση και τις συνεισφορές που μπορεί να γίνουν, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση με σωστό τρόπο, έτσι ώστε κάθε βουλευτής να μπορεί να συμβάλλει στο να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες και για τα κράτη και τις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μιλμπάο και κυρία Πατραωνέβες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γενικά συμφωνώ πολλά με πολλά πως επόθηκαν για την έκθεση αυτή. Επομένως δεν θέλω να επαναληφθώ. Θα ήθελα όμως καταρχήν να υπογραμμίσω ότι παραδοσιακά οι γυναίκες πάντοτε εργάζονταν στον κλάδο της ελιάς και για πάρα πολύ καιρό είχε έναν αόρατο ρόλο στον κλάδο αυτό. Σήμερα μιλάμε για 100.000 γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλίας. Το θέμα που συζητούμε σήμερα είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τον κλάδο της αλίας, αλλά αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ πιο συγκεκριμένα επικεντρωνόμαστε στην απασχολήση των γυναικών στον τομέα της αλίας που πάντοτε υπήρχε και αναγνωρίστηκε λίγο, Επίσης, αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποια βήματα προς την αναγνώριση και την ε, ε, αξιοποίηση του έργου των γυναικών, της δουλειάς των γυναικών σε αυτό το κλάδο και ερμηνεύω αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας ε, ως ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα εδώ να σας πω πως από την ακρόαση που κάναμε για το θέμα του ρόλου των γυναικών, εγώ είχα τη δυνατότητα να συναντήσω και αντιπροσώπους από τον κλάδο στην Πορτογαλία και να συζητήσω μαζί τους τα πιο σημαντικά θέματα σε σχέση με το θέμα αυτό που μας απασχολεί. Και ένα από τα σημαντικά θέματα που τονίστηκαν που υπογραμμίστηκαν έχει να κάνει με την αναγκαιότητα αναγνώρισης ε, και αξιοποίησης αυτού του ρόλου των γυναικών. την ε, ενεργοποίηση των ε, οργανισμών και των κρατών μελών και η ενεργοποίηση αυτή τι σημαίνει να υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση χωρίς ε, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να αναγνωριστεί ο ρόλος τους. Επίσης, μου τόνισαν θέματα που αφορούν ε, την ρύθμιση της δραστηριότητας των γυναικών στον τομέα της Ελίας, δηλαδή θέματα που αφορούν ε, θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλεια και τα εργατικά δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ρόλος που έχουν διαδραματίσει στον κλάδο και είπαμε ήταν λίγο αναγνωρισμένο, λίγο ορατός δεν είναι ένα θέμα μόνο κοινωνικής ορατότητας, αλλά έχει να κάνει και με την ασφάλεια των γυναικών στην εργασία και με κοινωνική στήριξη στην περίπτωση εγκυμοσύνης, συνταξιοδότησης, αρρώστιας κτλ. Επομένως πρέπει να ρυθμιστεί η εργασία των γυναικών στον κλάδο αυτό. Και Επίσης, έχουμε συζητήσει ότι όλες αυτές οι πτυχές θα είναι αντικείμενο καλύτερης υπεράσπισης όταν υπάρχει αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πράγματι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην το υδατοκαλλιέργεια έχει εργαστεί για να αυξήσει την προβολή των γυναικών που εργάζονται στην αλία και στην υδατοκαλλιέργεια. Επομένως, πρέπει να δούμε και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οργάνωσης αυτής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι επίσης σημαντικό να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το δίκτυο, το ακτέια. Αυτή τη στιγμή δεν ε, ε, υπάρχει εγγύηση για το ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί και αν ε, κατά κάποιο τρόπο δεν μπορέσουμε να εγγυθούμε αυτή η μεγάλη οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να αναπτύσσεται θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Αυτό η οργάνωση είναι πολύ σημαντική για την ανταλλαγή εμπειριών, για τη δημιουργία συμπράξεων και επίσης για την προώθηση της κατάρτισης των γυναικών για το ε, να μπορούν να ε, βρουν και άλλους τρόπους απασχόλησης και στον τομέα της αλίας και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι απαραίτητα για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που να ευνοούν την παραμονή των γυναικών στον κλάδο και την εξέλιξή τους. Γιατί αν δεν μπορέσουμε να εγγυηθούμε τη διατήρηση αυτού του ευρωπαϊκού δικτύου, τη συνέχιση της λειτουργίας τους, τότε αυτό θα σήμαινε παναχώρηση. Αυτά ήθελα να συνεισφέρω εγώ στη συζήτηση και ευχαριστώ και όσους ε, πήραν το λόγο για την εργασία τους και για την παρουσίασή τους. Ευχαριστώ κύριε Πατρεωνέβες. Κύριε Λιβέτη. Κλειβέτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να πω ότι για πρώτη φορά από το που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλέπω όχι μόνο ενδιαφέρον αλλά και πάθος ε, για το θέμα αυτό και πραγματικά αυτό είναι λογικό Γιατί όταν βλέπουμε να υπάρχει και ενδιαφέρον, ε, είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Εγώ προέρχομαι από την Ρουμανία και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει και εκεί ο κλάδος της αλίας ε, και έχουμε ίδια προβλήματα με τις γυναίκες. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν, όμως ως κοιόδης από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι Έχω παρατείνει κάποιες τροπολογίες όπου θέλω να αναφερθώ στην έλλειψη στατιστικών στοιχείων σε σχέση με το φύλλο, αυτό υπόθηκε, αλλά και κάποια μέτρα για να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να είναι αυτά αποσχολούμενες σε αυτό το τομέα και αναφέρουμε παραδείγματος χάρη στις μικροπιστώσεις που θα ήταν πολύ σημαντικές. Επίσης, η εγκαιότητα να αναπτυχθούν αυτές οι περιφέρειες όπου αυτή η δραστηριότητα είναι ο μόνος κλάδος που θα μπορούσε να επιφέρει εισόδημα ε, στους πολίτες ε, και δει στις γυναίκες. Υπάρχει και το γεγονό ότι στις ε, περιοχές αυτές βλέπουμε κάποια περιστατικά βίας κατά των γυναικών λόγω της ανέχειας, λόγω της ανεργίας. Βλέπουμε τέτοια φαινόμενα πιο συχνά σε σχέση με άλλους κλάδους, με το πόσο συμβαίνουν σε άλλους κλάδους. Επομένως, είναι σημαντικό για μας ε, να λάβουμε υπόψη και την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και οικονομικές σχέσεις ε, με άλλες χώρες ε, και σε αυτές τις χώρες ε, αυτή η δραστηριότητα είναι σημαντικό τμήμα της οικονομικής τους δραστηριότητας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τις γυναίκες και σε εκείνες τις χώρες στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και πάλι συγχαίρω τους δύο συγγητές. και θα υποστηρίξω την έκθεση αυτή με τροπολογίες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κλειβέτη. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Γκαμπρέλα Ιγκλόη από την ΓΑΜΑ Δελταμάρα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη μου παρέμβαση σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που με παρουσιάσατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την πρωτοβουλία αυτή του Κοινοβουλίου και την κοινή μάλιστα πρωτοβουλία των Επιτροπών Γυναικών και Αλληλείας και ιδιαίτερα την πολλή δουλειά που έκαναν οι δύο εισηγητές, η κυρία Γκαρσία Ιέρο και ο κύριος Ρωμέβα. Θα ήθελα να επιστρέψω και να αναφερθώ ξανά σε ορισμένα σημεία τα οποία ανέφεραν τα μέλη αυτή τη Επιτροπή, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία. Ε, μπορώ με αυτόν τον τρόπο να σα δώσω ορισμένε απαντήσει ή να επιβεβαιώσω τι ανησυχίε σα. Καταρχά, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία αναγνωρίζει την έμφυλη διάσταση. Έχει την οριζόντια αρχή της ε, μη διάκρισης και της ισότητας. Αυτό είναι έτσι μια πιο γενική δήλωση. Τι σημαίνει όμως την ουσία. Έχει σοβαρές επιπτώσεις σε δύο τομείς. Ο ένας είναι η εκπροσώπηση των δύο φύλων σε ε, οργανισμούς. Κάθε κράτος μέλος θα ε, πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, δηλαδή πρέπει και στην, στον προγραμματισμό να συμμετέχει και στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται σε όλα τα στάδια της λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου του Ταμείου αυτού. Έπειτα, η προώθηση των γυναικών σύμφωνα με τις αρχές αυτές αναγνωρίζεται ο ρόλος των γυναικών, των συζύγων, ε, των αλλιέων έτσι ώστε εκείνες να γίνουν ε, δικαιούχοι διαφόρων παροχών και με τις παροχές αυτές θα μπορέσουν να ε, αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες ή να βελτιώσουν τις υφισταμένες δεξιότητες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συμμετέχουν σε διάφορες ασκήσεις ανταλλαγής εμπειριών. Τώρα, να απαντήσω στην ε, κυρία Γερόκα σε ένα σχόλιο που έκανε για την ε, ε, σημασία της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Να σας πω ότι έχουμε κάτι τέτοιο, τον άξονα 4, ο οποίος αναγνωρίζεται ως το σημαντικότερο στατικό στοιχείο του MFF όσον αφορά την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν διατάξεις ε, κατά τις οποίες οι γυναίκες που είναι δικαιούχοι ε, συμμετέχουν ταυτόχρονα και στην εφαρμογή του προγράμματος. Και αυτό θα συνεχιστεί και στο επόμενο πρόγραμμα, με άλλη ονομασία όμως, ε, ανάπτυξη κοινοτήτων και τοπική ανάπτυξη. Ελπίζουμε, όμως, ελπίζουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του μέσου αυτού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Εγκλό και καλώς ήλθατε στην Επιτροπή αυτή. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τους εισηγητές το λόγο να ολοκληρώσουν. κυρία Γκαρσία η το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλες τις συναδέλφους ε, βουλευτές που πήραν το λόγο. Νομίζω ότι συμπίπτουν οι απόψεις μας και η ανάλυση που κάνουμε του θέματος, όπως επίσης και οι προτάσεις και οι τροπολογίες τις οποίες ενδεχομένως θα καταθέσουν, τις οποίες καλοδέχομαι. Όντως η έκθεση αυτή, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε μέχρι να βρεθεί εδώ που βρίσκεται, μπορεί τελικά να είναι τυχερή. Προσπαθήσαμε όλοι οι εισηγητές για τους διάφορους κανονισμούς να καταθέσουμε τροπολογίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες, είναι για την ισότητα των γυναικών, για να είναι πιο ορατή η εργασία των γυναικών, για να έχουν ε, τρόπους να εκπροσωπούνται περισσότερο, για να συμμετέχουν πιο πολύ, για να εκπαιδεύονται καλύτερα. Και έχουμε και τη μελετή την οποία εγώ παρουσίασε την παρουσίασα εγώ στην Επιτροπή για την οποία δυστυχώς δεν αισθάνθηκα πως δείξατε την ίδια ευαισθησία γιατί εμείς εδώ έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλία. Θα ήταν καλύτερο όλα αυτά να τα είχαμε κάνει στους κανονισμούς. Εκεί να ήμασταν πιο δεκτικοί. Γιατί βεβαίως έχουμε ένα ταμείο ε, έχουμε νέες ε, εκπαιδεύσεις, έχουμε μικροπιστώσεις, έχουμε νέες επιχειρηματίες, έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη, μιλάμε για άξονα 4, αλλά μόνο ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη την... Ε, και την δραστηριότητα των γυναικών στην αλληλεία. Μόνο ένα. Νομίζω λοιπόν πως είναι η κατάλληλη στιγμή να το προωθήσουμε και στους κανονισμούς, ανεξάρτητα με το ότι η έκθεση αυτή, που είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, κρούει ένα κόδωνα κινδύνου. Να δούμε δηλαδή εάν θα καταφέρουμε να έχουμε ένα δυναμικό τελικό αποτέλεσμα. Ακόμα υπάρχει χρόνος. Και επειδή είδα να υπάρχει ευαισθησία, το ίδιο είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχω καμία αμφιβολία. Επίσης, η Επιτροπή Αλληλείας, οι εισηγητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον τριμερή διάλογο, σίγουρα θα κάνουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα στοιχεία τα οποία είχαμε πει κάποτε πως θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός να ενταχθούν και στα δικά τους θέματα και αναγνωρίζω πως Έχουμε πολλές πρωτοβουλίες, έχουμε το πρόγραμμα Horizon και νομίζω ότι και οι γυναίκες ερευνητέ ε, σε θαλάσσια θέματα θα πρέπει να στηριχθούν. Και πρέπει να σας πω πως ε, δείχνουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μια μεγαλύτερη ευαισθησία, γιατί από το 2005 και μετά δεν είχαμε κάνει τίποτα και πέρασαν πολλά χρόνια. Είμαστε λοιπόν όλοι υπεύθυνοι. Πρέπει να σας πω, παρόλο που οι γυναίκες αυτές είναι σκορπισμένες, παρόλο που δεν φαίνονται, είναι 100.000 άνθρωποι που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα αυτού του κλάδου. Κάτι που πάντα μας ανησυχεί. Στην περιβαντολογική βιωσιμότητα της περιοχής τους. Στην οικονομική τους βιωσιμότητα, στην οικογενειακή τους βιωσιμότητα. Και είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος μένει εκτός της νομικής αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της υγειονομικής κάλυψης. Και αυτό βέβαια θα επηρεάσει και ε, τη συντάξη τους και τη δυνατότητα που θα έχουν ε, να πάρουν τα διάφορα επιδόματα μητρότητας. Σας καλώ λοιπόν, ό,τι δεν είχαμε συμπεριλάβει στις τροπολογίες, να τα τοποθετήσουμε τώρα εδώ στην έκθεση αυτή τη βδομάδα, έτσι ώστε, όπως είπε η Σάσκο Βιλμπάου, να μην έχουμε απλώς ένα στόχο, αλλά μια πραγματική δέσμευση. Γιατί την αρμοδιότητα ποιοι την έχουν. Για τη διαχείριση τα κράτη-μέλη και αυτόνομες περιφέρειες, αλλά για την επαλήθευση, για τον έλεγχο, για την πρόθεση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεύθυνη. Και ας εξετάσουμε εάν μπορούμε αυτά να τα εντάξουμε. Είναι μια έκκληση αλλά και μια απέτηση. Γιατί αν υπάρχει αυτή η ομοφωνία πως πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν το συμφωνούν αυτό οι δύο επιτροπές του Κοινοβουλίου, τότε θα πρέπει να φαίνεται και στους κανονισμούς, γιατί δεν θα έχουμε άλλη τέτοια ευκαιρία μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Και η έκθεση τι μας λέει. Πως θα μπορούσαμε να είμαστε σε, μια... σε ένα διαφορετικό σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Εγώ ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα έπρεπε να επαναλάβω τέτοια τέτοια επιχειρήματα στη ζωή μου, γιατί το έκανα παλιά, για τις γυναίκες που ε, προσέχουν τις οικογένειές τους, για τις νοικοκυρές, ε, για, τα, για τις εσωτερικές οικιακές βοηθούς. Ε, νομίζω πως υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και αυτή τη στιγμή μιλάμε για την αλία που αποτελούν έναν πυλώνα βασικό της οικονομίας της ζώνης τους. Και κλείνω με αυτό. Ζούμε σε συγκυρία κρίσης. Είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και θα πρέπει να βρούμε νέες πρωτοβουλίες. Και αυτό άκουσα από το δίκτυο γυναικών. Ήταν εκπληκτική η συμμετοχή. Και κάθε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία έρχονται να που είναι δυο λόγια. Μας είπαν, οι ενώσεις τους δεν έχουν οικονομικούς πόρους. Δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν ε, όσους συμμετέχουν σε ενώσεις τους. Δεν έχουν πόρους για να φτιάξουν μια σελίδα, μια ιστοσελίδα και να επικοινωνούν έτσι μεταξύ τους. Θα χρειαστεί λοιπόν να πρικοδοτηθούμε τα απολύτως απαραίτητα έτσι ώστε να τα καταφέρουν. Οι γυναίκες είναι πολυμήχανες. Γεννημένες επιχειρηματίες. Οπότε σίγουρα και στις περιοχές αυτές ό,τι και να προσφέρουμε ε, θα το χρησιμοποιήσουν. Και όταν ξεπεράσουμε την κρίση θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε καλύτερα την εργασία τους και ίσως τότε θα μπορούμε να συγχαρούμε λίλους πως τουλάχιστον κοινωνικά και νομικά αναγνωρίστηκε το έργο τους από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Thank you Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαρσία. Ο κύριος Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσω κι εγώ δύο Το πιο σημαντικό στοιχείο της συζήτησης αυτής είναι το θέμα της αναγνώρισης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν τη δουλειά των ανθρώπων αυτών και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι πρέπει να το κάνουμε, οφείλουμε να το κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να ε, δούμε που είναι το πρόβλημα και κατόπιν να το επιλύσουμε στα πλαίσια της συζήτηση που έχουμε τώρα αλλά και στον τριμερή διάλογο για το Ταμείο Αλίας θα εκμεταλλευτούμε ένα παράθυρο ευκαιρίας που μας δίνεται και θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε την οικονομική αλλά και την νομική αναγνώριση των γυναικών που δεν είναι ίσονο σημασία ζήτημα. Και κάτι ακόμα που δεν το είπαμε, αλλά νομίζω είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Όχι μόνο μιλάμε για τις γυναίκες ε, που δραστηριοποιούνται στις ελευτικέ δραστηριότητες αυτές καθ' αλλά και στις δραστηριότητες της θάλασσας. Γιατί μερικές φορές ε, ξεχνάμε ε, τις δραστηριότητες των γυναικών που μπορεί να απασχολούνται σε κάποιους τομείς που έχουν σχέση με τη θάλασσα και υπάρχει αντίκτυπο στις εργασίες τους στον ελευτικό τομέα. Επομένως, ε, όλο αυτό το θέμα μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε πολιτικό αλλά και θεσμικό επίπεδο για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το, το θέμα. Και με τη συνάδελφο, την κυρία Γκαρσία Ιέρο, θα απαντήσουμε σε όλα τα αιτήματα, γιατί αν και έχουμε περιορισμό ε, σε ό,τι αφορά τους ε, χαρακτήρες. Ε, όποια συνεισφορά θεωρούμε ότι βελτιώνει το κείμενο, από εμάς θα είναι απολύτως αποδεκτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές, τον κύριο Ρωμαβή και την κυρία Ιέρο. Και ευχαριστώ ένθερμα και την Επιτροπή την εκπρόσωπο από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Πάντοτε θέλουμε να συνεργασόμαστε μαζί σας. 4 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 22-23 Ιανουαρίου και προβλέπεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 4, πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπών. Εμείς ε, ε έχουμε